Υποφορία θα λάβει χώρα αύριο στις 12. Το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι μια στιγμή Α, ναι. το μέλλον της Συμφωνίας Ασφαλούς Λιμένα of υπό το φως της υπόθεσης NSA. Να σας ενημερώσω, αγαπητοί συνάδελφοι, πως η συζήτηση αυτή δεν ε, θα έχει την διαδικασία της μπλε κάρτας. Γι' αυτό και δεν θα γίνουν δεκτές ερωτήσεις. Να ξεκινήσουμε με τον κύριο Υπουργό εκ μέρους του Συμβουλίου. Έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, τους τελευταίους έξι μήνες ε, είδαμε ανησυχητικές διαρροές στα ΜΜΕ που αφορούν τα μυστικά προγράμματα παρακολούθησης ε, που επηρεάζουν τα προσωπικά δεδομένα και την ιδιωτική ζωή των Ευρωπαίων πολιτών. Η αποκάλυψη πληροφοριών για τα προγράμματα που ε, έχει η NSA, η Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας των ΗΠΑ, οπωσδήποτε εγείρει ανησυχίες. Ε, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα αντέδρασαν με διάφορους τρόπους. Βεβαίως ε, συστήσατε μια δική σας εξεταστική επιτροπή η οποία από ό,τι καταλαβαίνω σύντομα θα καταλήξει σε μια έκθεση. Επιπροσθέτως υπάρχει μια ομάδα εργασίας ad hoc για την προστασία των δεδομένων με τις ΕΠΑ για να εξετάσει το νομικό πλαίσιο για τις δραστηριότητες παρακολούθησης που αφορούν τους κατοίκους της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι πρόεδροι από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης της ομάδας αυτής εκτός αν πέρσι 27 Νοεμβρίου μια έκθεση. Επίσης η Κομισιόν δημοσίευσε μια ανακοίνωση τον Νοέμβριο για την ε, αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στις ροές ε, δεδομένων. Όσον αφορά το ζήτημα αυτό του ασφαλούς λιμένα είναι ένα ζήτημα της Κομισιόν καθώς πρόκειται περί απόφασης της Κομισιόν ως μέρος ε, των υποχρεώσεών της. Η Κομισιόν πρόσφατα εξέδωσε μια ανακοίνωση που απευθύνεται στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο για τη λειτουργία της απόφασης αυτής. Ως ένα πρώτο βήμα η Κομισιόν προγραμμάτισε μια συζήτηση εις βάθος μεταξύ εκπροσώπων των κρατών μελών στην ε, λεγόμενη Επιτροπή του άρθρου 31 αυτή θα είναι η αρχή της αναθεώρησης της λειτουργίας του συστήματος αυτού και αντιλαμβανόμαστε πως η διαδικασία αυτή θα περιλαμβάνει μια ανοιχτή διαβούλευση και συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η έκθεση της Ομάδας Εργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης ήπα ΕΕ, δείχνει πως η Αμερικανική νομοθεσία περιέχει κάποιες νομικές βάσεις που επιτρέπουν την συλλογή σε μεγάλη κλίμακα και την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που μεταφέρονται στις ήπα ΕΕ, ε, και εκεί πέρα υφίστανται επεξεργασία. Η απόφαση αυτή στο παράρτημα 1 προβλέπει πως μπορεί να περιοριστεί η αρχή της ιδιωτικής ζωής εάν κάτι τέτοιο δικαιολογείται από την εθνική ασφάλεια, το δημόσιο συμφέρον ή απαιτήσει των διοκτικών αρχών. Η Κομισιόν δηλώνει στην ανακοίνωσή της πως ενώ η κατεξαίρεση είναι επεξεργασία δεδομένων για σκοπούς εθνικής ασφάλειας αναγνωρίζεται η πρόσβαση η μαζική ε, από τις υπηρεσίες ε, πληροφοριών στα δεδομένα τα οποία πηγαίνουν στη ΣΥΠΑ στο πλαίσιο εμπορικών συναλλαγών δεν προβλεπόταν όταν ε, εγκρίθηκε το νομοθέτημα αυτό. Η ανακοίνωση της Κομισιόν έκανε 13 συστάσεις για να βελτιωθεί η λειτουργία του ασφαλούς λιμένα. Όσον αφορά την πρόσβαση από αρχές των ΙΠΑ σε δεδομένα που μεταφέρονται υπ' αυτόν τον τρόπο πρέπει να αναφέρουμε τρία στοιχεία πρώτα απ' όλα οι αρχές της αναλογικότητας και της αναγκαιότητας πρέπει να γίνονται σεβαστές αυτό σημαίνει να δούμε τις πιθανές διαφορές ε, ερμηνείας μεταξύ ΕΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης για το τι είναι αναγκαίο και αναλογικό ειδικά για την προστασία της εθνικής ασφάλειας επίσης συμβαίνει πως πρέπει να δούμε τις πιθανές διαφορές μεταχείρισης ε, Αμερικανών πολιτών και κατοίκων και μη Αμερικανών πολιτών. Την πιθανή, όπως είπα, διαφορετική μεταχείριση. Δεύτερον, η Κομισιόν εκφράζει ανησυχίες για το ότι κάποιες από τις δικλείδες ασφαλείας που προβλέπει η νομοθεσία της Αμερικής ισχύουν μόνο για πολίτες και μόνιμους κατοίκου νόμιμους κατοίκους ΗΠΑ. Η Κομισιόν έχει εκφράσει ανησυχία για αυτά. Υπάρχει ανάγκη ίσης μεταχείρισης μεταξύ κατοίκων Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών αναγνώριση εφαρμόσιμων δικαιωμάτων ε, για τους Ευρωπαίους πολίτες όπως και για τους Αμερικανούς και η ανάγκη να ενισχυθεί η αναλογικότητα και το κριτήριο της αναγκαιότητας για τη συλλογή αυτών των δεδομένων. Όπως ξέρετε στις ΕΠΑ αυτή τη στιγμή επανεξετάζεται η λειτουργία των προγραμμάτων παρακολούθησης και ελπίζουμε να ληφθούν υπόψη αυτά τα οποία ανέφερα. Το τρίτο που έθεσε η Κομισιόν είναι η ανάγκη μεγαλύτερης διαφάνειας για τα δεδομένα που έχουν μεταφερθεί στις ΕΠΑ σύμφωνα με την συμφωνία αυτή. Η έκθεση της ομάδας αναθεώ, ε, εξέτασης των τεχνολογιών κατασκοπίας ε, που συνέστησε ο πρόεδρος Ομπάμα έχει κάνει κάποιες ε, συστάσεις. Τώρα θα έρθουμε σε επαφή με τις Πολιτείες για να δούμε ακριβώς πώς θα αντιμετωπιστούν αυτά τα οποία αναφέρει η Κομισιόν στην ανακοίνωσή της. Ενώ το πίμαχο ζήτημα βεβαίω είναι οι πρακτικές της NSA, οι συστάσεις της Κομισιόν αναφέρουν και άλλες πτυχές της λειτουργίας και εφαρμογής ε, της Συμφωνίας Ασφαλώς Λεμένα. Θεωρούμε πως έτσι πρέπει να προχωρήσουμε. Πρόκειται για μια απόφαση της Κομισιόν που βασίζεται στην Οδηγία Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του 1995, οπότε θεωρούμε πως είναι αρμοδιότητα της Κομισιόν και όχι του Συμβουλίου να τροποποιήσει ή να ανακαλέσει την απόφαση αυτή. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, διακυβεύονται σημαντικά ζητήματα εδώ πέρα. Αφενός, όλες αυτές οι ανησυχίες για συλλογή πληροφοριών από τρίτη χώρα που την χάνει να είναι ο σημαντικότερος στρατηγικός μας εταίρος. Αφετέρου, πρέπει να λάβουμε μέτρα, να προστατεύσουμε το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή ε, των ανθρώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τελικά αυτό το ζήτημα μπορεί να λυθεί μόνο μέσω διαλόγου και άρα είναι δεκτές όλες οι ευκαιρίες για συζήτηση και ενθαρρύνουμε την Κομισιόν να συνεχίσει τον επικοδομητικό διάλογο με τις αρχές των ΙΠΑ επί των ε, συγκεκριμένων σημείων που ε, χρήζουν προσοχή. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Το λόγο έχει η Αντιπρόεδρος της Κομισιόν, κυρία Ρέντινγκ. Ευχαριστώ αγαπητά μέλη. Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε τις επιπτώσεις των αποκαλύψεων για την NSA το καλοκαίρι σε πολλές ε, περιστάσεις και περιπτώσεις και εδώ και στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Οι ανταλλαγές ήταν πολύ χρήσιμες και προσβλέπω ε, τα συμπεράσματα της ε, Επιτροπής Έρευνας της ΛΥΜΠΕ. Θα πρέπει να μιλάμε με ενιαία φωνή να προβάλλουμε νέα στάση έναντι των ΙΠΑ και η προστασία δεδομένων θα πρέπει να τύχει ε, σωστής αντιμετώπισης με βάση τις ανταλλαγές και συναντήσεις με τις αρχές των ΙΠΑ και τις ε, επισκέψεις μας στις ΙΠΑ, καθώς ε, και τη συνάντηση στην Επιτροπή Ad Hoc Ευρωπαϊκή Ένωση ΙΠΑ, τονίσαμε τις ανησυχίες μας και μιλήσαμε με μία φωνή από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Κοινοβουλίου. Και έτσι ακριβώς ε, αυτή η ενιαία φωνή δηλαδή εισπράχθηκε στις ΗΠΑ. Είπαμε προς τις ΕΠΑ ότι θα πρέπει να οικοδομήσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης στην διατλαντική σχέση και στη σχέση ανταλλαγής πληροφοριών, κάτι το οποίο έχει διαραγεί. Όπως ανέφερε και η Προεδρία, ο ασφαλής λιμένας είναι μια σημαντική συμφωνία και διευθέτηση σε αυτά τα πλαίσια. Ε, είναι ε, θέμα ευθύνης της Επιτροπής. Μιλάμε για διαβίβαση δεδομένων προς επιχειρήσεις των ΙΠΑ και στόχος αυτής της ε, συμφωνίας αρχικά του 2000 ήταν να διασφαλίσουμε τα δικαιώματά μας σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα με βάση και τα ευεργετήματα μεταφοράς δεδομένων προς επιχειρήσεις των ΗΠΑ, προς ε, αντιμετώπιση. Τώρα όμω υπάρχουν πολλές ε, ελλείψεις και προσπαθούμε να τις αντιμετωπίσουμε. Αναλύσαμε λοιπόν τη συμφωνία αυτή του ασφαλούς ε, λιμένα και στις 27 Νοεμβρίου ε, εκδώσαμε αυτό το συμπέρασμα και ίσως ο ασφαλής λιμένας να μην είναι και τόσο ασφαλής ε, διαχρονικά. Επειδή λοιπόν υπάρχει έλλειψη διαφάνειας από πλευράς ΙΠΑ, ορισμένες ε, επιχειρήσεις έμπρακτα δεν συμμορφώνονται με το πρόγραμμα αυτό όπως ε, είχε οριστεί. Αυτό έχει αρνητικές επιπτώσεις στα προσωπικά δικαιώματα και οδηγεί σε ένα συγκριτικό πλεονέκτημα ανταγωνισμού αυτών των επιχειρήσεων κατά των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που δρούν στην ίδια αγορά. Επίσης, διαβλέπουμε τους κινδύνους της συμφωνίας αυτής του ασφαλούς λιμένα, διότι οι αρχές ασφαλείας των ΗΠΑ έχουν πρόσβαση μέσα στα πλαίσια μιας ευρύτατης παρακολούθησης, ενώ η συμφωνία ε, κάνει λόγο για περιορισμένες πληροφορίες όταν ε, βασίζονται σε θέματα ε, εθνικής ασφαλείας, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την αρχή της αναλογικότητας και της αναγκαιότητας. Δεν μπορούμε να δεχτούμε συλλογή πληροφοριών για πρόσωπα εκεί που δεν υπάρχουν υποψίες. Αυτό δεν είναι ούτε αναγκαίο ούτε αναλογικό. Και κατέστησα σαφές τους Αμερικανούς ομολόγους ότι αυτό το θέμα θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε ικανοποιητικά αν θέλουμε να, να διασφαλίσουμε τη συνέχεια της Συμφωνίας Ασφαλούς ε, Λιμένα. Είπα, θα πρέπει να δεχτούν την διαφάνεια και εάν διαβιβάζονται αυτά τα στοιχεία στις ΕΠΑ δεν θα πρέπει να αναλύονται από την NSA. Ο στόχος Συμφωνίας Ασφαλούς Λιμένα ήταν να υπάρχει ένα υψηλότερο επίπεδο προστασίας από αυτό που προβλεπόταν από τον Εθνικό Νόμο των ΗΠΑ για να τηρηθούν οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές προστασίας προσωπικών δεδομένων. Άρα η Συμφωνία Ασφαλούς Λιμένα θα πρέπει να προστατεύει τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών κατά τη διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ. Θα πρέπει λοιπόν να ε, δούμε τη σωστή ε, λειτουργία της Συμφωνίας του Ασφαλούς Λιμένα και αναγνωρίζουμε 13 βασικά σημεία για την πραγματική προστασία δεδομένων σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και υποβάλαμε συγκεκριμένες συστάσεις σε τέσσερις βασικούς τομείς για βελτίωση, προσβελτίωση που θα πρέπει να τύχουν αποδοχής για τη διαφάνεια, για την, περίπτωση χρήσης ενδικών μέσων, πραγματική εφαρμογή και τον περιορισμό πρόσβασης από τις δημόσιες αρχές. Με αυτά τα 13 σημεία οι Αμερικανικές αρχές έχουν επιτάπητος έναν κατάλογο καθηκόντων και ελπίζω να μπορέσουν να βελτιώσουν τη συμφωνία αυτή. Θα γίνει μια πρώτη διερευνητική συνάντηση στις Βρυξέλλες ε, στο εγγύς μέλλον με τις αρχές των ΙΠΑ και το Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και η Επιτροπή Εμπορίου των ΗΠΑ, με τις οποίες έχω συνδιαλλαγή, μίλησαν για βελτίωση της Συμφωνίας Ασφαλούς Λιμένα και εξαιρέσεις μόνο όταν υπάρχουν θέματα εθνικής ασφάλειας που θα πρέπει να ερμηνευτούν συσταλτικά. Δηλαδή να χρησιμοποιηθεί αυτό το δικαίωμα όταν είναι αναγκαίο και αναλογικό ε, όπως έχει οριστεί εκ των προτέρων. Η ανακοίνωσή μας για την οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνη στη ροή δεδομένων δείχνει ότι θα πρέπει μέσα στα πλαίσια του έτους να προβλεφθούν ε, μέτρα, αντισταθμιστικά μέτρα και μετά θα ε, αναθεωρήσουμε την λειτουργία της Συμφωνίας Ασφαλούς, ασφαλούς Λιμένα με βάση την όλη διαδικασία εξέτασης μέσα στα πλαίσια μιας ανοιχτής διαβούλευσης και συζήτησης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αγαπητά μέλη, θα πρέπει ο ασφαλής ε, λιμένας να γίνει ακόμα πιο ασφαλής. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να γίνει αναθεώρηση διαβίβασης προσωπικών δεδομένων. Θα πρέπει να οριστούν ε, σαφείς κανόνες όταν διαβιβάζονται στοιχεία και την χάνουν εξέτασης. Πρόκειται για ένα πρόκριμα για την νομική ασφάλεια ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις. Γι' αυτό θα ήθελα να συγχαρώ όσους εργάστηκαν για την αναθεώρηση της προστασίας δεδομένων πολύ σκληρά. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέστησε σαφές, σαφή την θέληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να ασκήσουμε πίεση προς το Συμβούλιο να επιταχύνει τις εργασίες έτσι ώστε να αρχίσουν οι διαβουλεύσεις και να συναυθεί μια συμφωνία με βάση τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και είμαι ευγνώμων προς την Ελληνική Προεδρία γιατί την επόμενη εβδομάδα προβλέπεται μια άτυπη, συνάντηση η οποία προβλέπει αυτό το θέμα προς συζήτηση. Ευχαριστούμε κυρία Ρέντινγκ. Πριν αρχίσω τη ζήτηση, υπενθυμίζω, συνάδελφοι, ότι κατά τη ζήτηση αυτή δεν προβλέπονται ούτε μπλε κάρτες, ούτε η διαδικασία προσέλκυσης της προσοχής του Προέδρου. Η συζήτηση, λοιπόν, θα περιοριστεί σε έναν εκπρόσωπο πολιτική ομάδα. Λοιπόν, ο αντιπρόεδρος του ΕΛΚ, κύριος Μάνφρεντ Βέμπερ. Τρία λεπτά. Ε, κύριε Αντιπρόεδρε, κύριε Εκπρόσωπο του Συμβουλίου, κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής. Η συζήτηση καθιστά σαφέ σήμερα ότι πρέπει να επιμείνουμε ως Κοινοβούλιο. Θέλουμε οπωσδήποτε ζήτηση για το NSA να παραμείνει ζωντανή. Είναι μήνυμα προ του πολίτε στην Ευρώπη ότι ασχολούμεθα με το θέμα αυτό, αλλά και προ του ε, φίλου μα στην Αμερική. Το πολιτικό πλαίσιο είναι σαφέ. Η NSA, με βάση αυτό που μάθαμε και οι διαστάσει αυτών που μάθαμε, ήταν αδιανόητε για πολλού από εμά και μπορούμε να συγκρίνουμε με την Κίνα και τη Ρωσία. Αλλά τώρα έχουμε να κάνουμε με τους Αμερικανούς φίλους μας. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση. Οι πρώτες απαντήσεις ήταν σωστές πολιτικές και μετά η Κομισιόν και η Επιτροπός μας κατέστησε σαφές προς την Washington και, αλλά, τι επιθυμούμε, αλλά και η Επιτροπή Έρευνας πρέπει οπωσδήποτε να καταστήσει σαφές όπως και τα κράτη-μέλη τι επιθυμούμε. Πρέπει να απαντήσουμε με, στο επίπεδο που θέλουμε ως Ευρώπη και πρέπει να δούμε και νομοθετικά το θέμα. Αυτή είναι η πρόκληση. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα αλλιώς θα είναι κατά αυτής της απόφασης για τον ασφαλή λιμένα. Πρέπει να ασκήσουμε πίεση για τα τίθεται το ερώτημα εάν και κατά πόσο οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι ασφαλής λιμένας ή εάν δεν είναι πλέον ασφαλής λιμένας. Διότι η αρχή του ασφαλούς λιμένα ήταν αρχή της αγοράς η αμοιβέ, ο αμοιβαίος σεβασμός των ε, αρχών του, της προστασίας των δεδομένων. Γι' αυτό θέλουμε να επεξεργαστούμε το δικό μας δίκαιο για την προστασία των δεδομένων και δεν είναι δυνατόν να το εφαρμόσουμε μόνο για τις ε, ευρωπαϊκές εταιρείες εάν δεν ε, ισχύει ουσιαστικά για όλες τις εταιρείες ο ασφαλής λιμένας. Θέλουμε λοιπόν όλες οι υπηρεσίες που χορηγούνται στην Ευρώπη να ε, συμμορφούνται προς το ευρωπαϊκό δίκαιο. Γι' αυτό πρέπει να εξετάσουμε λοιπόν αυτό το θέμα αυτό. Και κυρίως γιατί είμαστε στην αρχή της ε, ψηφιοποίησης. Τα επόμενα χρόνια και δεκαετίες θα διαπιστώσουμε ότι θα αλλάξει εντελώς η ζωή μας. Και ο δεύτερος λόγος για τον οποίο θέλουμε να καταργηθεί αυτή η συμφωνία είναι ότι ελπίζουμε ότι έτσι η Ευρώπη θα καταλάβει ότι οι Ευρωπαίοι αντιμετωπίζουν σοβαρά την κατάσταση αυτά στα πλαίσια της τροποποίησης της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης ότι πρέπει η Washington να αντιμετωπίσει εκ νέου το θέμα. Αυτό διαφορετικά δεν θα αποδεχθούμε στο μέλλον οι πολίτες μας ή αν θέλετε οι καταναλωτές να είναι πρώτης και τέτοιες κατηγορίας να είναι δηλαδή σε άλλο επίπεδο για το θέμα του επίπεδου προσθέσεων των δεδομένων Ευρωπαίοι από τους Αμερικανούς και θέλω να υποστηρίξω σαφώς την Κομισιόν ότι πρέπει οι πολίτες μας και οι εταιρείε μας να έχουν τη δυνατότητα στην Ευρώπη να απαιτήσουν αυτά τα, να κάνουν αυτές τις απαιτήσει και η Ευρωπα... το Ευρωπαϊκό Ελληνικό Κόμμα θέλει εταιρική σχέση με τις ΗΠΑ και με αυτόν τον τρόπο, με την κατάργηση αυτής της συμφωνίας, θέλουμε να δημιουργήσουμε νέα βάση για αυτήν την εταιρική σχέση. Ε, να είναι μια εταιρική σχέση που να αξίζει αυτό το όνομα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δήμπα. Και τώρα από πλευράς των σοσιαλιστών, ο κύριος Κλωτ Μωράες. Τρία λεπτά μετά από αυτή την ομιλία να πω ότι αν υπάρχει συμβολική αλλά και ουσιώδη σημασία της έρευνα του Κοινοβουλίου κατά αυτή της μαζικής παρακολούθησης είναι η εξέταση του θέματος του ασφαλούς λιμένα, γιατί αφορά τους πολίτες μας, τα προσωπικά τους δεδομένα, αφορά και εμπορικά και βιομηχανικά και ε, οικονομικά ε, συμφέροντα και λειτουργίε. Είναι λοιπόν συμβολικό των προβλημάτων που έχουμε με τη μεταφορά των δεδομένων, το πρόβλημα εμπιστοσύνη που έχουμε μεταξύ ε, Ένωση και ΗΠΑ. Και είναι συμβολικό του τι πρέπει να διορθώσουμε. Ο ασφαλή λιμένα, από πολλέ απόψει, έχει γίνει σύμβολο της κατάσταση που αντιμετωπίζουμε και των καθηκόντων που έχουμε ενώπιόν μα. Αυτή η έρευνα και το σχέδιο εκθεσής μου μαζί με τους κοιόδης φυσικά που είναι εδώ παρόντες και με βάση το έγγραφο εργασίας του Axel Βόστ όλη αυτή η ε, σημαντική δουλειά που έχουμε κάνει στους τελευταίους μήνες κατέληξε στην σύσταση να αναστείλουμε αυτή τη συμφωνία ούτω ώστε να διασφαλίσουμε τη δημιουργία ενός άλλου μηχανισμού που να καταγράφει το υψηλότερο επίπεδο προστασίας δεδομένων που έχουμε εμείς στην Ένωση. Ο κύριος Βέμπερ πολύ σωστά τα είπε. Δεν είναι να τον έχουμε δύο κατηγορίες πολιτών, δύο κατηγορίες επιχειρήσεων. Είναι απαράδεκτο. Τι λέμε λοιπόν για τον ασφαλή λιμένα που είναι τόσο και συμβολικό και συγκεκριμένο. Πρώτα αναφερόμαστε στις αδυναμίες και στην έλλειψη πληροφόρησης. Γιατί είδαμε στην Εξεταστική Επιτροπή ότι ορισμένες εταιρείε που δεν συμμορφούνται παραμένουν ε, να αναφέρονται στο site του FTC ως ε, συμμορφούμενες. Και δεν έχουμε και επαρκή μηχανισμό προσφυγής, ούτως ώστε να υπάρχει δυνατότητα απεύθυνση στη δικαιοσύνη και να μπορούν και οι εταιρείε να απευθύνουν στη δικαιοσύνη. Αυτές είναι οι δυναμίε που διαπιστώσαμε. Τα στοιχεία που συλλέγονται από τους πολίτες τη Ένωσης μεταφέρονται με ιδιαίτερα δύναμες εγγυήσει. Μεταφέρονται στι ΗΠΑ. Γνωρίζοντα ότι στι ΗΠΑ είναι χαμηλότερα τα επίπεδα προστασία των δεδομένων. Ο ασφαλή λιμένα όπω έχει τώρα δεν προσφέρει, δεν εγγυάται στου πολίτε μα καμία προστασία έναντι ε, αιτήσεων από ε, το NSA για πληροφορίε με βάση την, ε, τον, νόμο, τον πατριωτικό νόμο στις ΗΠΑ. Και ξέρουμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ηλεκτρονική παρακολούθηση από πλευρά από των ΗΠΑ που θεωρούμε ότι παραβιάζει τις αρχές της συμφωνία. Η Κομισιόν ήδη, ήδη έχει αναγνωρίσει τις σοβαρέ αδυναμίες του ασφαλούς λιμένα. Αλλά αυτό μπορεί να μην αρκέσει η διαδικασία δεν έχει καμία δυνατότητα όπω είναι αυτή τη στιγμή να εφαρμόζεται. Και γι' αυτό δεν την παίρνουν στα σοβαρά οι ΗΠΑ. Θα ήθελα λοιπόν να πω στην ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνούμε και μιλάμε με μια φωνή προ την Ουάσιγκτον. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι ο ασφαλή λιμένας έχει συμβολική και πρακτική σημασία. Πρέπει να διορθωθεί η κατάσταση για να δημιουργηθεί εκ νέου εμπιστοσύνη στι σχέσεις και για να έχει πραγματική έννοια ούτω ώστε ο κανονισμό για προστασία των δεδομένων να παίξει ουσιαστικά το ρόλο του στη σχέση μα με τι ΗΠΑ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία, η κυρία Σοφία Ινφελτ από πλευρά ε, των Φιλελευθέρων. Παρακαλώ, δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, Σα ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για τα λόγια σα και την πρότασή Σα. Είναι καλή αλλά ειλικρινά όχι αρκετή. Το ξέραμε εδώ και χρόνια Πολλοί προ πω πως η συμφωνία αυτή ήταν λανθασμένη και ήταν απλά συμβολική. Δεν παρέχει καμία προστασία στους Ευρωπαίους πολίτες, παρά μόνο νομική κάλυψη στις εταιρείε που επεξεργάζονται δεδομένα στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη και γνωρίζουν πώς παραβιάζουν το ευρωπαϊκό δίκαιο. Και επειδή δεν θέμε να τους δημιουργήσουμε προβλήματα, ανεχτήκαμε την κατάσταση. Για πολλά χρόνια και ζητήσαμε από την Κομισιόν επανειλημμένα να ε, βρει μια λύση, αλλά δεν έκανε τίποτα. Μάλιστα, αυτή η περίφημη αξιολόγηση της ε, συμφωνίας ή της συνεννόησης αυτής, νομίζω έγινε δύο χρόνια μετά την προθεσμία. Γιατί λοιπόν να δώσουμε και άλλο χρόνο στην Κομισιόν και στη ΣΥΠΑ να βρουν μια λύση. Ξέρουμε ποιο είναι το πρόβλημα, ξέρουμε πώς δεν λειτουργεί και ειλικρινά έχω αρχίσει να χάνω την υπομονή μου με τις εταιρείε αυτές. Γιατί όπως είπα εδώ και πολλά χρόνια ανοιχτήκαμε την κατάσταση για να τους δώσουμε μια ευκαιρία. Και τι κάνουν σε αντάλλαγμα ασκούν πιέσεις για να αποδυναμώσουν την προστασία των δεδομένων. Από ότι ε, εγώ θεωρώ πω πρέπει σήμερα να αναστείλουμε τη συμφωνία για να κινητοποιηθεί επιτέλου και η Κομισιόν και η Αμερικανική κυβέρνηση και οι εταιρείε για να αρχίσουν να ψάχνουν μια σοβαρή λύση. Γιατί έχει φτάσει η ώρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο και η Κομισιόν να υπερασπιστούν τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών, οι οποίοι πρέπει να προηγούνται των διεθνών σχέσεων και των επιχειρηματικών συμφερόντων. Και αυτό το λέω πραγματικά πόνο ψυχής γιατί είμαι φιλελεύθεροι. Αλλά πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Οπότε κυρία Επίτροπε, αναμένω από την Κομισιόν να αναστείλει την συμφωνία σήμερα και να έχουμε επαρκείς λύσεις. Προσεχώς, πριν από τις εκλογές. Σας ευχαριστώ. Για 1,5 λεπτό ο κύριος Άλμπρεχτ ε, για λογαριασμό των Πρασίνων. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε κύριε Επίτροπε, κύριε Υφυπουργέ, κύριε συνάδελφοι. Η αποκαλύψη του Edward Snowden έδειξαν ότι χρειαζόμαστε καλύτερη προστασία για τα προσωπικά δεδομένα. Ο τρόπο με τον οποίο ε, οι μεγάλε επιχείρησει στον τομέα αυτό και οι υπηρεσίε προφοριών ε, ε, εισβάλλουν στον προσωπικό μα χώρο είναι απαράδεκτο. Αλλά παρά το ότι εκατομμύρια πολίτε και καταναλωτέ δημοσίου διαμαρτύρονται γι' αυτό, ούτε μία κυβέρνηση τη Ένωση δεν έχει κάνει κάτι για να το σταματήσει. Και εδώ δεν ακούω να κάνει κανεί κάτι, να ε, προσπαθεί να κάνει κάτι συγκεκριμένο. Αντίθετα, η φωνή του Google, ο Eric Schmidt, λέει ότι η προστασία των δεδομένων είναι ανώμαλη κατάσταση και θέλει να σταματήσει. Οι επιχειρήσεις του Silicon Valley έκαναν επιτυχημένες προσπάθειες λόμπι κατά οποιασδήποτε ρύθμιση της προστασίας δεδομένων στην Washington. Εδώ στην Ευρώπη μας αγνούν. Χρησιμοποιώντας την συμφωνία για τον ασφαλή λιμένα, εισβάλλουν και αποφεύγουν οποιαδήποτε, ε, οποιοδήποτε περιορισμό τη Ευρωπαϊκή αρχέ, Αγαπητοί συνάδελφοι, να σταματήσουν όλα αυτά. Το Κοινοβούλιο έχει τη δυνατότητα να το κάνει. Έχουμε επιμείνει στην ε, υιοθέτηση ε, ενό ενιαίου νομοθετήματο για την προστασία των ευρωπαϊκών δεδομένων εδώ και δύο χρόνια. Όμω οι συνάδελφοι στο Συμβούλιο των Υπουργών πηγαίνουν γύρω-γύρω χωρίς να έχουν καμία διάθεση να καταλήξουν ούτως ώστε να υπάρξει ουσιώδης προστασία και οι μεγάλες επιχειρήσεις ε, δεδομένων στη Silicon Valley τι λένε ευχαριστώ πολύ ενώ οι πολίτες της Ένωσης και οι καταναλωτές χάνουν κάθε εμπιστοσύνη στις ε, δυνατότητε των κυβερνήσεών μα να υποστηρίξουν και να προστατεύσουν μερικά από τα πιο θεμελιώδη δικαιώματά μα. Εάν δεν σταματήσει η καταστρατήγηση των ευρωπαϊκών κανόνων από τι ε, εταιρείε των ΗΠΑ μέσω νομοθεσίας, ενιαία νομοθεσίας του κανονισμού αυτού και ασκώντα πίεση στι ΗΠΑ, Καταργώντα ε, την απόφαση για τον ασφαλισμένο, όχι μόνο θα χάσουμε κυριαρχία ως Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θα χάσουμε και τους ψηφοφόρου, οι οποίοι δεν θα έρθουν να ψηφίσουν, γιατί δεν περιμένουν να προστατεύσουμε τα συμφέροντα και τα δικαιώματά του. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η κυρία Κορνέλια Έρνστ ε, της Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Ε, ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, τι πρέπει να κάνουμε με τις σχέσεις μας με τις επα. Θέλουμε να είμαστε κυρίαρχοι απέναντι στις επα. Να καταγγείλουμε την ε, συμφωνία ή θα κάνουμε πάλι τους ε, καλούς και οι άλλοι θα κάνουν μεγάλο αδερφό και θα γελάνε μαζί μας. Η συμφωνία αυτή επί της αρχής είναι καλή, αλλά στην πράξη είναι φάρσα. Δεν έχει απομείνει κανένα δικαίωμα με το πατριωτικό νόμο τον ΗΠΑ. Αυτά εδώ πέρα δεν αξίζουν το χαρτί που έχουν γραφτεί καν. Έτσι, καμία επιχείρηση δεν μπορεί να διωχθεί για οτιδήποτε έχει κάνει. Κανένας έλεγχος, καμία προσφυγή. Εντάξει, μπορεί να έχετε καλές προθέσεις, αλλά δεν φτάνουν αυτά. Και πάμε σε λάθος δρόμο. Χρειαζόμαστε υψηλή προστασία των προσωπικών δεδομένων, υποχρεωτική για όλες τις επιχειρήσεις, αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου, όπως και να το πείτε, πρέπει να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο, μια συμφωνία με τη ΣΥΠΑ η οποία θα είναι δεσμευτική. Και βεβαίως μπλοκάρεται οποιαδήποτε τέτοια συμφωνία και δεν παραχωρούν ούτε ένα εκατοστό, ούτε μια σπιθαμή. Και επιφυλάσσονται το δικαιώματό τους να παρακολουθούν τους Ευρωπαίους πολίτες. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να μας αντιμετωπίζουν έτσι σαν θυράματα. Τι να πω. Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 ε, μπορεί να καταγγελθεί αυτή η συμφωνία αν δεν εφαρμόζεται. Αναμένω λοιπόν από την Κομισιόν και για τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων πάνω από 500 εκατομμυρίων πολιτών να το κάνει αυτό. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Τζαβέλα για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα είμαι προκλητική. Αλλά ε, ας έρθουμε και στον πραγματικό κόσμο. Οι εθνικές κυβερνήσεις και οι υπηρεσίες ασφαλείας στόχο έχουν να διαφυλάξουν ε, την ευημερία των πολιτών τους. Και πρέπει να έχουμε κατά νου πως ο λόγος για τον οποίο απολαμβάνουμε αυτή την υψηλή ποιότητα ασφάλειας ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και της ΕΠΑ είναι λόγω ακριβώς των μηχανισμών αυτών ασφαλείας. Δεν λέω κατά κανένα τρόπο πως ε, τα βασικά δικαιώματα των πολιτών πρέπει να παραβιάζονται. Μάλιστα, τα προγράμματα αυτά διασφαλίζουν ακριβώς το αντίθετο, την προστασία των πολιτών και της ιδιωτικής ζωής τους. Κυρίε και κύριοι, θα ήθελα να υπενθυμίσω την τρομοκρατική επίθεση στη Βοστόνη πέρσι στο Μαραθώνιο. Εάν δεν υπήρχε επιτήρηση, αν δεν υπήρχαν οι κάμερες, οι τρομοκράτες δεν θα είχαν βρεθεί ποτέ. Η Ευρώπη είναι παράδειγμα φιλελεύθερης κοινοβουλευτικής δημοκρατίας και δεν πρέπει να θεωρούμε πώς ε, πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα ζητήματα αυτά μέσω της νομοθεσίας. Σας ευχαριστώ κυρία Τζαβέλα. Ε, προς την κυρία Σόφη Ινετφέλντ να υπενθυμίσω πως δεν υπάρχει μπλε κάρτα σε αυτό το θέμα. Για τους μη εγγεγραμμένους, ο κύριος Μάρτιν Έρενχάουζερ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Θυμάμαι τη δεκαετία του 90. Τότε υπήρχε μεγάλη εμπορευματοποίηση και υπήρχε και μια μεγάλη αντίδραση που ήθελε να υπάρχει ένα ελεύθερο και μεταοικονομικό ίντερνετ. Ήταν ουτοπία και από αυτήν την ουτοπία δεν έχει μείνει τίποτα. Αντίθετα, αντί για ουτοπία έχουμε δυστοπία. Πρέπει να πω λοιπόν ότι οι μηχανισμοί προστασίας που έχουμε δεν έχουν καμία επίδραση. Και ούτε τα σκάνδαλα και ούτε οι μεταρρυθμίσεις δεν προχωρούν. Ούτε τα σκάνδαλα δεν βοηθάνε να υπάρξει αλλαγή. Αυτό έχει να κάνει ε, από το γεγονός ότι εν μέρη από την Κομισιόν και εν μέρη από τα κράτη-μέλη μπλοκάρονται. Χρειαζόμαστε ενιαία δράση, χρειαζόμαστε μεταρρυθμίσεις στον τομέα της ε, διακυβέρνησης του ίντερνετ, ε, για τις ε, οικονομικές λειτουργίες του ίντερνετ και θα πρέπει να υπάρχει και καλύτερος έλεγχος των μυστικών υπηρεσιών. Αν τα έχουμε όλα αυτά, τότε αυτό που συζητάμε σήμερα δεν έχουν καμία έννοια. Δεν τις θέλουμε αύριο αυτές μεταρρυθμίσεις, αλλά σήμερα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η κυρία Ρέντιν για να ε, κλείσουμε τη συζήτηση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητά μέλη. Ε, κατανόησα απόλυτα και έλαβα το μήνυμά σας. Και εσείς κατανοείτε ότι όπως ζητήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αναλύσαμε το καθεστώς ασφαλούς λιμένα και με βάση την εργασία της ομάδας ad hoc και τις συζητήσεις με τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις είδαμε που υπάρχουν ελλείψεις και συμφωνώ για αυτά που είπατε ως προς αυτές τις ελλείψεις. Αυτά είναι τα συμπεράσματα τα οποία είναι ίδια με τα δικά μας. Και με βάση αυτά τα συμπεράσματα η Ευρωπαϊκή Επίτροπη υπέβαλε 13 συγκεκριμένες συστάσεις που σχετίζονται με όλες τις ε, πτυχές του προγράμματος, δηλαδή διαφάνεια, χρησιμοποίηση ένδικων μέσων και ε, ενδυνάμωση της ασφάλειας, ενίσχυση της ασφάλειας. Αυτά τα 13 αιτήματα συστάσεις βρίσκονται στην πλευρά των Αμερικανών θα πρέπει να τις αναγνωρίσουν αυτές τις συστάσεις καθώς και τις ανησυχίες μας. Η συζήτηση σήμερα θα μας βοηθήσει να προχωρήσουμε, να κάνουμε ένα βήμα προς τα εμπρός. Και βεβαίως ε, μέχρι το καλοκαίρι του 2014 θα πρέπει να δούμε πού θα πρέπει να καταφύγουμε σε ένδικα μέσα και το Διευθυντήριο των Επιτρόπων θα αποφασίσει από αυτόν. Και θα ήθελα να σας τονίσω ότι θα αποτανθώ στο Διευθυντήριο και θα αναφερθώ στη συζήτηση που είχαμε σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ την Επίτροπο και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Κούρκουλα. Εξ Συμβουλίου. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, ο μόνος τρόπος να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα που συζητάμε είναι ο διάλογος με τη ΣΥΠΑ. Σύμφωνα με την συμφωνία αυτή, η αρμοδιότητα αυτή ανήκει στην Κομισιόν και θα ήθελα να ζητήσω η Κομισιόν να έχει τον χρόνο και την εμπιστοσύνη να το κάνει. Όπως και το Σώμα, έτσι και το Συμβούλιο θα παρακολουθήσει το τι κάνει η Κομισιόν σε σχέση με αυτή την απόφαση. Πολλές από τις ανησυχίες που ακούστηκαν ε, είναι σωστές, αλλά βεβαίως πρέπει να επιτρέψουμε στην Κομισιόν και στις αρχές των ΗΠΑ να έχουν αρκετό χρόνο στη διάθεσή τους για να δουν αυτά τα ζητήματα. Σε λίγους μήνες ε, η ομάδα τεχνολογιών κατασκοπίας και επικοινωνιών υπέβαλε την έκθεση της ε, και η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το ίδιο. Πρέπει τώρα να επιτρέψουμε να υπάρξει αρκετός χρόνος για να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα αυτά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Έκλεισε και αυτό το θέμα. Περνάμε στο επόμενο. δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής για την ε, ηθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς πώληση. ήθελα λοιπόν και πάλι να δώσω τον λόγο στον κύριο Υπουργό